Συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είχε διακοπή 28 του 2009. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε να πω δύο λόγια. Όπως γνωρίζετε, πριν από δέκα ημέρες, ο Λέχ Κασίνσκι, πρόεδρος της Πολωνίας, κύρωσε τη συνθήκη της Λισαβόνας. Και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 η έκκλησή μας προ ε- πάσα χώρα και προσπάθησε κατεύθυνση για ένα απόλυτο μορατόριο στις εκτελέσει θενατικής ποινή σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ. Και τώρα προχωρούμε στην ε, έγκριση των πρακτικών.